witam państwa otwieram posiedzenie Καλημέρα σα. Άρχεται η συνεδρίαση. Η κυρία Χέρτσοκ, Καλημέρα σε όλου, κύριε Πρόεδρε. Χτε έγινε μια συζήτηση επί του προπολογισμού και ήταν σαφέ κατά τη διάρκεια τη συζήτηση πως η έκθεση της Επιτροπής Ήτρε δεν είχε πάει στις υπηρεσίες. Το ελέγξαμε αυτό. Είχε αποσταλεί σωστά η έκθεση, οπότε πιθανώς κάτι έγινε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αλλά σημασία δεν έχει να βρούμε τι ακριβώς συνέβη, αλλά το σημαντικότερο είναι ε, η έκθεσή μας που αποτέλεσε την ε, βάση του τριμερούς διαλόγου και βεβαίως ε, είχε και κάποιες διαφορές σε σχέση με το αρχικό έγγραφο και πρέπει να πάει στο Συμβούλιο. Οπότε την έφερα μαζί μου και σας παρακαλώ να τη διαβιβάσετε στο Συμβούλιο για να είμαστε σίγουροι πώς θα φτάσει εγκαίρως η έκθεση η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε αυτό το οποίο θέλετε από εμάς. Καταλάβατε. Ε, είναι φανταστική η αρχή της σημερινής συζήτησης. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι κοινή συζήτηση για την σύνοδο κορυφή των G20 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε δηλώσει του Συμβουλίου και της Επιτροπής ε, για την συνάντηση της 11 η και 12ης Νοεμβρίου και για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 28 και 29 Οκτωβρίου. Επιπλέον έχουμε την έκθεση